Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, einen schönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Καλημέρα σας, αγαπητοί ε, συνάδελφοι. Αρχίζει η συνεδρίαση. Πρώτο, πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η κοινή συζήτηση για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Σερβίας. Υπάρχει μια σύσταση Κατσίνσκ για την, το σύμφωνο σταθεροποίησης της Ευρωπαϊκής και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής ε, κοινότητες και της Σερβία και μία συμφωνία, μία δήλωση μάλλον του Συμβουλίου για τη Επιτροπή. Πρώτο ε, ε, ομιλητής, ο κ. Κατζίνο, ε, εισηγητή, τέσσερα λεπτά έχει τη διάθεσή σας. Ευχαριστώ, Σιλβάνα. Κύριε Επίτροπε, η Βελγική Βελική Προεδρία, εκπρόσωποι της Βελικής ε, Προεδρίας, αγαπητοί συνάδελφοι, η Συμφωνία Σταθεροποίησης υπεγράφει τον Απρίλιο του 2008 και έχει τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή το 2010. Το 2008 το Σερβικό Κοινοβούλιο ήταν το πρώτο που κύρωσε αυτή τη συμφωνία. Στην ουσία γίνεται λόγος για το πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο συνεργασίας. Χωρίς τη διαδικασία κύρωσης δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί η διαδικασία ολοκλήρωσης της ένταξης. Το θέμα αυτό δεν ευρέθη στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από τη διαδικασία κυρώσεων, διότι υπήρχε ανεπαρκή συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουκοσλαβία. Προς το παρόν, αρκετές χώρες έχουν κυρώσει την συμφωνία και θα ήθελα να καλέσω και τις υπόλοιπες να κάνουν το ίδιο. Στη συνέχεια θα αποστείλουμε ένα στεναρό μήνυμα προς τη Σερβία για να συνεχίσει αυτές τις προσπάθειες. Το ψήφισμα το οποίο θα ψηφιστεί αύριο, η πρόταση ψηφίσματος, θα πρέπει να αποστείλει ένα μήνυμα υποστήριξης προς την Σερβία. Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα είχε απομονωθεί η Σερβία και αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Στο παρελθόν είδαμε μία πολιτικοποίηση της κατάστασης in situ θα πρέπει η Σερβία να ενστερνιστεί τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προβεί στις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις. Έχουν υπάρξει και θετικές εξελίξεις. Η Σερβία θα δεχτεί ένα ψήφισμα, δέχτηκε το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών το 2010 για το Κωσυφοπαίδιο και επίσης δεν υπάρχει υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Οι νέοι Σέρβοι έχουν πλέον την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και στον, στην τριτογενή, στην ε, ανώτερη εκπαίδευση. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι υπάρχουν ε, δύο φυγόδικοι οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθερα. Ο Ράτκο Μλάντιτς είναι πρόσφυγας θεωρείται πρόσφυγας και θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τις αρχές της Σερβίας που δέχονται αυτή τη συνεργασία και θα θέλαμε ο κύριος εισαγγελέα, οι γνωματεύσει του κυρίου του επικεφαλής εισαγγελέα να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τη Σερβία. Ήρθε η ώρα έτσι ώστε η Σερβία να κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός. Δεν μπορεί να θεωρηθεί υποψήφια χώρα πριν αποδείξει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουκοσλαβία. Αυτό αφορά την έκδοση των εγκληματιών πολέμου κυρίως. Επίσης, έχουν γίνει, έχουν επέλθει αλλαγές και στα πλαίσια των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό το βλέπουμε και στις σχέσεις μεταξύ Κροατίας και Σερβίας και δόθη νέα όθηση για μία μακροχρόνια συμφιλίωση στην περιοχή. Η Σερβία θα πρέπει να κρατήσει επικοδομητική στάση και έναντι του πεδίου και αυτό είναι αναγκαίο έτσι ώστε ολόκληρη η περιοχή να μπορέσει να προοδεύσει. Το ίδιο ισχύει και ως προς τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Σερβίας και Βοσνίας Ερζεγοβίνης για να προωθηθούν οι διαπραγματεύσεις για αυτή την προσέγγιση των δύο χωρών. Η Υπουργός Γιώρη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που είμαι πάλι εδώ ως εκπρόσωπος ε, του Συμβουλίου της Προεδρίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ότι θα με θεωρήσετε πρώην μέλος ε, αυτού του Κοινοβουλίου. Και βεβαίως η Ουγγρική Προεδρία θα είναι φιλική Προεδρία ε, με μεγάλη χαρά θα συνεργαστώ με όλους σας κατά τη διάρκεια ε, του εξαμήνου αυτής ε, της Προεδρίας. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω στην δική μου την μητρική γλώσσα. Είναι πολύ μεγάλο προνόμιο που μπορώ να λάβω μέρος σε αυτή τη συζήτηση μετά την οποία θα ψηφίσετε για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Σερβίας. Θα ήθελα επίσης να υποφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να απευθύνω ευχαριστίες στον κύριο Κατσίνα, τον εισηγητή της, του Κοινοβουλίου που ετοίμασε μια πραγματικά εξαίρετη εισήγηση και χαιρετίζω το ψήφισμα επίσης σχετικά με την πρόοδο της Σερβίας. Όπως και άλλες χώρες της περιοχής, η προοπτική του να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεθάρρυνε την Σερβία για να κάνει πρόοδους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος στον δρόμο προς την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ε, συμφωνία ε, συσφίγγει ακόμα περισσότερο τις στενές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Σερβία και τοποθετεί τις σχέσεις αυτές σε μια βάση νομική, συμβατική, δημιουργεί μια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών και ενισχύει τις διμερείς οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στα δύο μέρη και θα ωφελήσει τόσο τη Σερβία όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία επίσης θα προωθήσει μέτρα της ε, Σερβίας ε, για την ανάπτυξη μιας αγοράς, ε, μιας οικονομίας της αγοράς που να λειτουργεί πλήρως και θα θέσει τα θεμέλια για μελλοντική ενισχυμένη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Σερβία σε πολλούς τομείς όπως το οργανωμένο έγκλημα, την, το παράνομο διασυνοριακό εμπόριο και τα θέματα του περιβάλλοντος. Το Συμβούλιο έχει αρχίσει στις 14 Ιουλίου 2010 την διαδικασία επικύρωσης. 11 κράτη-μέλη επικύρωσαν τη συμφωνία μέχρι τώρα και συμπεριλαμβανομένης και της Ουγγαρίας και ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσουν όλα τα άλλα κράτη-μέλη σε ένα προσεχές μέλλον. Το Συμβούλιο θα ήταν ικανοποιημένο αν μπορούσε η συμφωνία αυτή να τεθεί σε ισχύ στο τέλος του 2011 το αργότερο. Αυτό θα σήμαινε ότι η Σερβία θα έχει φιλόδοξες σχέσεις με την Ένωση σε μια εποχή όπου η διαδικασία ένταξης θα αποκτήσει πλήρη όθηση. Ελπίζουμε ότι θα υποστηρίξετε τη διαδικασία αυτή και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχει ψηφίσει ομόφωνα υπέρ της συμφωνίας αυτής. Η Σερβία υπέβαλε το αίτημα για προσχώρηση τον Δεκέμβριο 2009 ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις ευρωπαϊκές της προσδοκίες. Το Συμβούλιο θα γνωμοδοτήσει το δεύτερο εξάμεινο του 2011 γνωρίζουμε όλοι ότι η ενταξιακή διαδικασία της Σερβίας θα είναι ωφέλιμη για τη Σερβία. Υπάρχουν όμως μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν στο, σχετικά με το κράτος δικαίου, σχετικά με την ενίσχυση της δομής της δικαιοσύνης και στη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία. Όπως λέχθηκε στην εισήγηση του κυρίου Κάτσιν, η ενταξιακή διαδικασία θα λάβει υπόψη αυτές τις εξελίξεις και μερικές από τις εξελίξεις αυτές είναι πραγματικά σημαντικές. Θα ήθελα να υποφεληθώ της ευκαιρίας αυτής για να μιλήσω για τα ιστορικά μέτρα που έλαβε η Σερβία για να συνεργαστεί με τους γείτονές της. Ακόμη και τις ε, διαβουλεύσεις που είχε με την Ένωση το Ιούλιο του 2000 ε, που ε, ήταν, προκάλεσαν ένα ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών για την συνεργασία με το Κωσυφοπαίδιο και τα μέτρα που έλαβε η κυρία Άστον αυτή η συνεργασία και ο διάλογος ανάμεσα στο Κωσυφοπέδιο και στην Σερβία θα επιτρέψει στις δύο χώρες αυτές να, να πλησιάσουν τον στόχο της ένταξης. Πρέπει να είναι αξιόπιστη η διαδικασία η ενταξιακή και η διαδικασία διεύρυνσης. Έχουμε όλα τα μέσα για το σκοπό αυτό. Αν μπορούμε να κλείσουμε τις διαπραγματεύσει ενταξιακές με την Κροατία, αυτό θα στείλει ένα μήνυμα θετικό στη Σερβία και στις χάλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που θα ήθελαν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, το 2011 θα είναι σημαντική χρονιά για την Σερβία με προκλήσεις αλλά και με ευκαιρίες. Χαιρετίζω και επικροτώ αυτή την συμφωνία και τις ευκαιρίες που προσφέρει και που θα μας επιτρέψουμε να οικοδομήσουμε ένα κοινό μέλλον σε μια κοινή Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπος Φίλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να βρίσκομαι εδώ και να απευθύνομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα σε ό,τι αφορά την ε, ψηφοφορία αυτή, την έγκριση της ε, Συμφωνία Σταθεροποίηση και Σύνδεση με τη Σερβία. Θα ήθελα επίση να εκφράσω τι ευχαριστίε μου προ τον εισηγητή για τα θέματα τη Σερβία, τον κύριο Κάτσιν, για την έκθεση αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Ενσωμάτωση τη Σερβία. Συμφωνία σταθεροποίηση και Σύνδεσης είναι πολύ σημαντικό βήμα για τη Σερβία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και βασικό στόχος τη Συμφωνία αυτής είναι να προλιάνει το έδαφος για την περαιτέρω ευρωπαϊκή ε, ε, ενοποίηση και τις μεταρρυθμίσεις και να προετοιμάσει την τη Σερβία για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το σημαντικό ορόσημο θα αποτελέσει ένα κίνητρο, μια ενθάρρυνση για τη Σερβία για να ανανεώσει τις προσπάθειές της για την επανασυμφιλίωση στην περιοχή. Η Συμφωνία Σταθεροποίηση και Σύνδεση ε, δημιουργεί ένα συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο μέσα το Συμβούλιο SAA και την Επιτροπή αυτή ένα νέο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο σε επίπεδο υποεπιτροπών που καλύπτουν εκτενώς τα πιο, τους πιο πολλούς τομείς των ευρωπαϊκών πολιτικών και εννοείται ότι δημιουργεί επίσης ένα συγκεκριμένο σώμα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της, κοινής, και της Σερβίας, την κοινή κοινοβουλευτική, μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή. Δημιουργείται λοιπόν ε, ε, μια ζώνη ελευθέρου εμπορίου και προβλέπεται η σταδιακή προσχώρηση στην εσωτερική αγορά το οποίο θα έχει όφελος διπλό και προς τη Σερβία και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και για την Κεντρική Ευρώπη τη διαδικασία την δεκαετία του 1990 θα δώσει μια όθηση η συμφωνία αυτή στην ε, σερβική αγορά και θα συνδράμει θα βοηθήσει τη Σερβία να κινηθεί προς μια εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά. Τα ωφέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτήν την συμφωνία αυτή είναι εξίσου σημαντικά. Η σερβική αγορά ανοίγει πλέον για τους Ευρωπαίους εξάγωγείς γιατί οι υψηλοί δασμοί σταδιακά θα εξαλειφθούν με εξαίρεση κάποια πολύ ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα σταδιακά ενσωματώνοντας τη Σερβία στην εσωτερική αγορά θα γίνουν πιο προβλέψιμοι οι όροι για τους επενδυτές και οι κανόνες σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και τον ανταγωνισμό θα εναρμονιστούν με αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ίδιο θα συμβεί και με τα πρότυπα σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Η αγορά δημοσίων συμβάσεων επίσης στη Σερβία σταδιακά θα ανοίξει προς τους Ευρωπαίους. Επίσης ε, υπάρχουν και άλλα πλεονεκτήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θα διευκολυνθεί η συνεργασία σε τομείς δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, τις μεταφορές, τα τελωνία και αυτά είναι μόνο ενδεικτικά παραδείγματα. Άρα θα συμβάλλει στην μεγαλύτερη αξιοπιστία και την πιο ε, αποτελεσματική διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής στην περιοχή. Τέλος, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η Σερβία είχε προετοιμαστεί για την ε, ε, ενδιάμεση συμφωνία η οποία τέθηκε σε ισχύ το Φεβρουάριο του 2010, αλλά την οποία ουσιαστικά είχε μερικά εφαρμόσει η Σερβία από τον Απρίλιο του 2008. Η Σερβία έχει δημιουργήσει λοιπόν πολλά θετικά, έχει σημειώσει πολλά θετικά παραδείγματα από την απόφαση του 2010 να ξεκινήσουν ε, οι συμφωνίες, η επικύρωση μάλλον της συμφωνίας, εννέα είναι τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν επικυρώσει τη Συμφωνία σταθεροποίηση και σύνδεση και άλλα δύο έχουν εγκρίνει κοινοβουλευτικά τη συμφωνία αυτή. Και η συμφωνία αυτή ε, καλύπτει όλο το εύρος του πολιτικού φάσματος. Γι' αυτό λοιπόν θα ακολουθήσει και επικύρωση και από άλλες ε, χώρες μέλη. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να ολοκληρώσω επικεντρώνοντας ε, στο ψήφισμα, το σχέδιο ψηφίσματος σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ένταξη της Σερβίας, σε ό,τι αφορά και την ε, πολιτική συζήτηση, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κάτσιν. Η έκθεση αποστέλει ένα μήνυμα θετικό, ένα θετικό μήνυμα και προς τις δύο κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή Προπτική της Σερβίας και ένα μήνυμα προσδοκίας σε ό,τι αφορά και το παρελθόν της Σερβίας και το μέλλον της για την ευρωπαϊκή προοπτική. Και αυτό είναι ιδιαίτερα έγκαιρο σε ό,τι αφορά την ε, προετοιμασία της εξέτασης της ε, αίτησης ε, υποψηφιότητας Ευρωπαϊκής, της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρσι παρευρέθησα στο και οι σερβικές αρχές πρέπει να σας πω ότι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να απαντήσουν σε ό,τι αφορά το ρηματολόγιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με θαρρύνει η έγκριση από την, Ευρωπαϊκή, από την Σερβική Κυβέρνηση ενός σχεδίου δράσης, το οποίο θα αποτελέσει ένα follow-up τη έκθεση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύσει τις απαντήσεις προς το ερωτηματολόγιο και τα μέτρα που έχουν λάβει οι σερβικές αρχές τους επόμενους μήνες προκειμένου να ολοκληρώσει την ε, αξιολόγησή της με απότερο σκοπό να εκδώσει μια γνωμοδότηση στο δεύτερο ήμιση του 2011. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως είπε και ο Ούγκρος συνάδελφος, ε, το 2011 θα είναι σημαντικό έτος για τη Σερβία, ένα έτος ε, σημαντικών προκλήσεων αλλά και ένα έτος σημαντικών ευκαιριών. Έχει προλιανθεί πλέον το έδαφος και οι στόχοι είναι γνωστοί. Εξαρτάται ωστόσο από τη Σερβία να ακολουθήσει το μονοπάτι που χάραξε και να πληρώσει τα κριτήρια που έχουν τεθεί, να ε, επαναδεσμευθεί στην διαδικασία διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι βέβαιος ότι με την κοινή μας ε, υποστήριξη η Σερβία θα συνεχίσει να κάνει τις σωστές ευρωπαϊκές επιλογές και να προχωρήσει σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες ενσωμάτωσης. Αυτό θα αποστείλει θετικό μήνυμα σε όλη την περιοχή, μια χρονική στιγμή όπου χρειάζεται να επιβεβαιωθεί η ευρωπαϊκή πρόπτικη για να ενισχυθεί και η ανάπτυξη αλλά και η ειρήνη στην περιοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε, Πρό... κύριε Πίτροπε, λέει η Πρόεδρος. Και να περάσουμε τώρα στους ομιλητές εξ ονόματος των ομάδων για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δύο λεπτά, ο κύριος Σόφλιν, έχετε το λόγο. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κάτσιν και νομίζω ότι η Σερβία επιτέλους αποφάσισε ότι διαβλέπει ένα ευρωπαϊκό μέλλον για την ίδια. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το καλύτερο σημείο εκκίνησης. Η αποφασιστικότητα της Σερβίας έχει άμεση σχέση με τους κλειδονισμούς την τελευταία 20 ετία. Δηλαδή ε, τον βομβαρδισμό του 1999, τον Σλόμπονταν Μιλόσεβις, τη βία, τις μαφίες και μία ιδιαίτερα τραυματική ιστορία. Γι' αυτό θεωρούμε ότι επιτύχαμε μία πολύ στεναρή νίκη για σταθερότητα και σταθεροποίηση. Στην περιοχή θα πρέπει ο Ράτκο Μλάντιτς να προσαχθεί στη Χάγη και να αναγνωριστεί και το κοσυφοπέδιο. Πρόκειται για ψυχολογικά ε, σύνορα, ας το πούμε, ή ορόσημα, διότι ο Μλάδης την χάνει υποστήριξης από ένα ε, τμήμα της σερβικής ε, επικράτειας. Επίσης, θα πρέπει να ασχοληθούμε με την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, το σύστημα δικαιοσύνης, την οικονομία της αγοράς και ένα άνοιγμα προς, ε, ως προς το παρελθόν της Σερβίας, δηλαδή να ανοίξουν τα εθνικά αρχεία. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μία δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση. Το δέχεται γενικότερα η κοινωνία και υπάρχουν και οι τεχνικές προδιαγραφές. Πιστεύω ότι το φθινόπωρο η Σερβία θα θεωρηθεί υποψήφια χώρα. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ε, μελλοντικό αυτό πλαίσιο. Θα ήθελα να καλωσορίσω έναν προσκαλεσμένο που παρακολουθεί τη συζήτησή μας, τον κύριο Προσιλαντέτσιτς,